Ευχαριστώ. Κατά. Ένας. Αποχές. Α, δύο κατά. Αποχές εγκρίνονται. Η τροπολογία δύο τώρα. Ο εισηγητής επίσης είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Ευχαριστώ. κατά. Τρεις, τέσσερις. Αποχές εγκρίνεται και αυτή. Έχουμε τώρα για την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία ή Κολέγιο μια τροπολογία για την απελευθέρωση ορισμένων κοντιλίων και η τροπολογία μας είναι η αρχική διατύπωση ή όπως λέμε εδώ initial wording, όχι των σοσιαλιστών, η αρχική διατύπωση. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος άλλος είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ του initial wording. Ευχαριστώ κατά. Οι σοσιαλιστές και οι γκουε. Αποχές μία. Οι περισσότεροι υπέρ της initial wording που εγκρίνεται. Τώρα τα σχόλια των πιλωτικών υπηρεματικών δράσεων και βαστικών εδώ να μιλήσει ο εισηγητής νομίζω. Οι συντονιστές το συζήτησαν εχθές και θα μας πει τώρα ο εισηγητής πώς έχει η διαπραγμάτευση, αν μπορούμε να τα ψηφίσουμε όλα μαζί ή όχι. Η συθονία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολλά τα κείμενα εδώ πέρα και έχω λάβει ένα αίτημα χωριστής, ξεχωριστής ε, ψηφοφορίας ε, για την τροπολογία που σχετίζεται με το Φόρουμ Κοινωνίας των Πολιτών Ευρωπαϊκή Ένωση Ρωσία στη γραμμή 190406, αν δεν κάνω λάθος, είναι στη σελίδα 13, και 32 σε αυτά που έχετε μπροστά σας και η χωριστή ψηφοφορία είναι στην πρώτη παράγραφο των παρατηρήσεων και αφορά την τρίτη πρόταση που έχει ως εξής. Το φόρουμ θα οργανωθεί στο περιθώριο της των διετών Συνόδων Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας. Και το αίτημα είναι να ψηφιστεί χωριστά αυτή η πρόταση, αλλά εγώ προτείνω να ψηφίσουμε υπέρ. Ευχαριστώ. Αν κατάλαβα καλά, είναι η μόνη ψηφοφορία που είναι χωριστή. Δεν ζητάει κανένα άλλο για κανένα άλλο σημείο χωριστή ψηφοφορία. Δεν σας πιέζω για κάτι τέτοιο. Αντίθετα, απλώς θέλω να καταλάβω σωστά. Για να μην χάσουμε τίποτα μέσα στην ταχύτητα. Και να μην να μείνει δυσαρεστημένα κάποια πολιτική ομάδα. Λοιπόν, ψηφίζουμε καταρχήν την παρατήρηση αυτή. Είμαστε στη σελίδα 31 του φακέλου αυτού. Αλλά το σχόλιο είναι στην σελίδα 32, πάνω-πάνω. Πρόκειται για ένα πιλωτικό σχέδιο για το Φόρουμ, την Κοινωνία των Πολιτών Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας. Και έχουμε την εξής φράση. Η φράση που ψηφίζεται χωριστά είναι η φράση που ανέφερε η Σιδονία. The form would be organized in the fringe of the biannual EU-Russia summits. Το φόρουμ θα οργανωθεί στο πλαίσιο της διετούς Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας. Η συγκέντρια είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ αυτής της φράσης. Υπέρ αυτής της φράσης. Ηλεκτρονική ψηφοφορία Ελπίζω να έχετε τις κάρτες σας. Νομίζω ότι είμαστε 50-50. Όχι, όχι. Θα, θα ψηφίσουμε με το χέρι. Σηκώστε το χέρι παρακαλώ, όσοι είναι υπέρ. Κοσιμία ψήφι υπέρ. Κατά. Λιγότερες είναι ούτως ή άλλως. Πολύ λιγότερες. Δεδομένων των παρόντων, έχουμε μεγαλύτερη κινητοποίηση της δεξιάς από την αριστερά. 21 ψήφι υπέρ, 14 κατά. Όποιος κινητοποιείται κερδίζει. Όσοι δουλεύουν περισσότερο κερδίζουν από αυτούς που κάθονται. Το υπόλοιπο το ψηφίζουμε on block. Όλο μαζί, υπέρ, ευχαριστώ, κατά, δύο ψήφοι κατά, αποχές, δεν υπάρχουν. Υιοθετείτε. Μπράβο στην εισηγήτρια. δια πάντα είναι δύσκολη υπόθεση. Αλλά τα ψηφίσαμε όλα. Έχουμε αυτές τις ε, επιπλέον τροπολογίες που αναφέραμε το πρωί, συν την τροπολογία των σοσιαλιστών για τους νέους ίδιους πόρους. Έχουμε όμως και άλλες ψηφοφορίες. Την ε, ψηφοφορία της έκθεσης Ματέρα, που είναι τέσσερις ουσιαστικά εκθέσεις, αλλά οι ίδιες ε, τροπολογίες εμφανίζονται κάθε φορά Έχετε την, ε, τον κατάλογο ψηφοφορία για το, τις τροπολογίες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο κινητοποίηση για την Παγκοσμιοποίηση. Στην παράγραφο 5 έχουμε μια τροπολογία, την υπαριθμό 1 του κυρίου Άλβαρο και Χάγκλουντ. Η συγγήτρια είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Όλοι. Εκτός από τους συντάκτες και την ομάδα τους. Απορρίπτεται. Επομένως, να ψηφίσουμε τώρα την τροπολογία 2. Νταρντέν και Γκριλιέ. Η συγκέντρια είναι πάλι κατά. Ποιο είναι υπέρ. Οι σοσιαλιστές. Και οι πράσινοι. ποιο είναι κατά. Πλειοψηφία. Απορρίπτεται. Α, ξέχασα τις αποχές. Αποχές. Η Γκουε. Χάρτον κτλ. Τροπολογία 3. Άλβαρο και Χάγκλουντ. Με προφορική τροπολογία της εισηγήτριας που την έχετε γραπτός. Την οποία δέχονται οι συντάχτες. Η εισηγήτρια υπέρ λοιπόν τη τροπολογία. Ψήφι υπέρ. Κατά. Κύριος Μποκρός. Αποχές των σοσιαλιστών και των πράσινων και της Γκουε. Χα. δεν έχει να πείτε τίποτα για αυτό το θέμα. Δηλαδή, κλείνει το στόμα της η Γκουε μπροστά στην τροπολογία Άλβαρο. Τελική ψηφοφορία, υπέρ. Κατά. Αποχές. Ευχαριστώ. Υιοθετούνται και οι τέσσερις εκθέσεις. Συγχαρητήρια κυρία Ματέρα. Τώρα, τι μας μένει. οι μεταφορές των πιστώσεων. Κύριε Σούριαν, τις μεταφορές του κυρίου Σούριαν τις είχαμε ψηφίσει. Υπάρχουν οι μεταφορές που αφορούν την έκθεση Ματέρα. Θα μπορούσαμε να τις ψηφίσουμε όλες μαζί αυτές τις μεταφορές. Ναι, θα μπορούσαμε. Υπέρ, είμαι υπέρ. Λοιπόν, όλες μαζί οι μεταφορές του κυρίου Σουριάν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ναι, τα ίδια. Ναι, λογικό, λογικό. Τώρα, μεταφορά 28, κύριε Σιγητά. Είστε υπέρ, μάλιστα. Μεταφορά 28, και τις 3 ε, και την 58 και την 53 μαζί. Είστε σύμφωνοι και τις τρεις μαζί. Όχι. Όχι, συγκητής. Για την 53, αν είναι δυνατόν, θα ήθελα να αναβληθεί η ψηφοφορία. Καλά. Ψηφίζουμε λοιπόν μαζί την 28 και την 52 και το 53 αναβάλλεται. Λοιπόν, κύριε Χάρτουγκ, δεν γίνεται να τις ψηφίσουμε χωριστά. Βεβαίως, βεβαίως. μόνο. Λοιπόν, ψηφίζουμε την 28, τη μεταφορά 28, υπέρ. Υπέρ, μόνο την 28. Κα, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα η 52, η 52 μόνη της υπέρ. υπέρ. Κατά. Αποχές. Μία αποχή. Και η 53 είπαμε αναβάλλεται για άλλη φορά. Λοιπόν, τότε τελειώσαμε και τις μεταφορές του Λάσλο Σουριάν. Τώρα έχει φύγει ο εισηγητής, αλλά... αλλά μπορώ να τον αντικαταστήσω εγώ, εκτός αν θέλει κανείς άλλος να το κάνει. Έχω εδώ τις οδηγίες του εισηγητή κυρίου Μάγκα. Τρεις αιτήσει μεταφορών για τα άλλα όργανα. Πρώτα για το δικαστήριο. Το δικαστήριο λοιπόν μεταφορά ενός εκατομμυρίου από την θέση των αμοιβών στη θέση άλλων αναγκών διοικητικών που ανταποκρίνονται στην πληρωμή πρόσθετων προσελελημένων υπαλλήλων. Ο διοικητής είναι υπέρ. Ποιος άλλος είναι υπέρ. Ευχαριστώ, κατά. Ευχαριστώ, αποχές. Μία αποχή. Εγκρίνεται. Μετά, άλλη μεταφορά της Επιτροπής των Περιφερειών. Με το άρθρο 47. Είναι απλό μια αλλαγή του οργανογράμματός της, δεν, δεν έχει επιπτώσει στον προϋπολογισμό. Χρειάζεται μεταφορά, αλλά χωρίς επιπτώσεις. Φυσικά ο συγκεκριτής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ? Ευχαριστώ, κατά, ένας. Αποχές. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. Τέλος. Πάλι μεταφορά για την Επιτροπή των Περιφερειών. υπέρ της μετεκπαίδευσης των μελών των υπαλλήλων της Επιτροπής των Περιφερειών επειδή υπήρξε πλεόνασμα, περίσευμα στο κέντρο εκεί στο μελικό σταθμό της Επιτροπής των Περιφερειών. Περίσευμα. Παίρνουν το ψωμί από το στόμα των παιδιών και το δίνουν στους γεροντότερους. Μπορούμε λοιπόν να τους έχουμε εμπιστοσύνη νομίζω για την καλή χρήση των χρημάτων τους. Η συγκήτηση είναι λοιπόν υπέρ και εγώ είμαι υπέρ. Ποιος άλλος είναι υπέρ. Θα ευχαριστώ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελείωσαν οι μεταφορές, τελείωσαν οι ψηφοφορίες, τελείωσε και η συνεδρίασή μας. Είναι μεσημέρι, δουλεύουμε πολύ γρήγορα, ευτυχώς διότι η διάσκεψη των Προέδρων μας ε, δημιουργεί και υπερορίες λοιπόν. Υπενθυμίζω ότι θα ξαναειδωθούμε στην Επιτροπή μας την Πέμπτη το απόγευμα ή δυνατόν τη αιτήση ορισμένων συντονιστών και συντονιστριών από τους σημαντικότερους μάλιστα ήδη από τις δύο, δύο dès 14 14h. Bon. Από τι 2. Για ψηφοφορία και με τις κάρτες σα. ε, γιατί θα γίνουν ηλεκτρονικά οι ψηφοφορίες. Όχι πολλές, αλλά είναι πιο εύκολο έτσι. Λοιπόν, με τις κάρτες. Μέχρι τότε θα επεξεργαστούμε τις πρόσθετε τροπολογίες το απόγευμα και μόλις γνωρίζω την ακριβή ώρα της διάσκεψης των Προέδρων, τότε διήν φάτερον ούτε η διάσκεψη των Προέδρων θα γίνει χωρίς να προσκαλέσει αντιπροσώπους μας και τότε μπορούμε να οργανώσουμε τη δουλειά μας όπως θέλουμε. Αυτό θα ήταν περίεργο βέβαια, αλλά θα μπορούσαμε έτσι να οργανωθούμε όπως θέλουμε. Είτε, λέγω, η διάσκεψη των Προέδρων θέλει να ξανασυζητήσει τον προπολογισμό με εκπροσώπους μας, οπότε Ανάλογα με την ώρα θα σας προτείνω συντονιστές πριν την ώρα εκείνη. Ας πούμε, εκτός αν γίνει στις 7 η διάσκεψη των Προέδρων, οπότε εμείς θα συνεδριάσουμε μετά. Άρα κανονικά πριν, πριν. Και βέβαια πριν τις ψηφοφορίες της Μίνι Ολομέλειας της Πέμπτης και πριν την κομπού των 2 η ώρα. Λίγη συνεδρίαση.